Voilà, Καθίστε παρακαλώ για να περάσουμε στην ψηφοφορία. Αρχίζουμε με την πρώτη ψηφοφορία. Είναι η έκθεση στο Γιανόφ. Ενιαία ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Πατράων Εύες. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Σάζερ. Επίσης ονομαστική ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση Σάζερ. Και εδώ έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτη έκθεση Σάζερ. Και εδώ έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ.